της κυρίας Λούνατσεκ για την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωσυφοπεδίου. Κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πίτροπε, συνάδελφοι. Ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ε, επιφορτισμένη με αυτό το θέμα, θα ήθελα πριν μπω στις ε, λεπτομέρειες της συμφωνίας να μιλήσω για τον ε, Ιμπραχή Μολτόβα που κέρδισε το βραβείο Σαχάροφ ε, το 1998, ε, που πέθανε πριν από 10 χρόνια, το 2006. Είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας του, κοσφο, του Κοσφοπεδίου, ένας μεγάλος ηγέτης των Αλβανών Κοσοβάρων και θα ήθελα να τον τιμήσουμε στην αρχή της συζήτησής μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοσφοπέδιο, η Συμφωνία ε, Σύνδεση και Σταθεροποίηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε μεταξύ του Οκτωβρίου του 2013 και του Μάιο του 2014. Ε, μονογράφηκε τον Ιούλιο του 2014. Το Συμβούλιο συμφώνησε να υπογραφεί στις 22 Οκτωβρίου του 2015 και υπογράφτηκε εδώ στο Στρασβούργο στις 27 Οκτωβρίου από την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη από εσά, κύριε Χάν, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Πρωθυπουργό Ιζα Μουστάφα του Κοσμοπεδίου και τον Υπουργό Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ε, Μπεκίμ Τσολάκου. Τώρα, ε, η Εθνοσυνέλευση του Κοσμοπεδίου στι 2 Νοεμβρίου 2015 το επικύρωσε αυτό το κείμενο και σήμερα, ε, μάλλον αύριο, εμεί θα ε, ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχεία μπορεί να τεθεί σε ισχύ. Είναι μια ιστορική στιγμή για το κοσφοπέδιο αυτή. Γιατί για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοσφοπέδιο θα έχουν συμβατικές σχέσεις. Είναι η πρώτη ε, προσπάθεια, επίσημη προσπάθεια για να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοσφοπέδιο. Βεβαίως ε, χρειάστηκε χρόνος, γιατί το κοσφοπέδιο είναι μια νέα χώρα. Η ανεξαρτησία ε, έλαβε χώρα πριν από 8 χρόνια και χρειάστηκε χρόνο στο Συμβούλιο χρόνο στο Συμβούλιο. Όμω, πεντε πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο, έχουν δώσει τη συνένεσή του. και αυτό είναι μεγάλο βήμα προ τα εμπρό. και θα ήθελα να παροτρύνω αυτά τα κράτη να αναγνωρίσουν το κοσφοπέδιο. Κάποιε από τι χώρε έχουν υπουργού οι οποίοι επισκέπτονται το κοσφοπέδιο, συναντώνται με αξιωματούχους κυβέρνηση. Σα παρακαλώ λοιπόν, κάντε τα απαραίτητα βήματα, αναγνωρίστε το κοσφοπέδιο. Κοσφοπέδιο είναι η νεαρότερη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν κάνει κακό, δεν βλάπτει, απλώ βοηθάει από του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία είναι και σταθεροποίηση. Τι είναι ακριβώ. Για πρώτη φορά εξασφαλίζει σημαντικέ σχέσει. Έχει, εξασφαλίζει έντονο πολιτικό διάλογο, νέε μορφέ συνεργασία, καλύπτει πολλοί αριθμούς τομείς, ε, ενισχύει τι δημοκρατικέ αρχέ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και ένα πλαίσιο για συνεργασία σε τομεί όπω η εκπαίδευση, η ενέργεια, περιβάλλον, δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσει και πολλοί πολλοί άλλοι τομεί. Επίσης, ε, μιλάει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και είναι ένα τεράστιο κίνητρο για την εφαρμογή και θεσμοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Γιατί το κοσμοπέδιο χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνηση θα πρέπει να τις κάνει. Επίσης δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις ταυτόχρονα ε, για καλή διακυβέρνηση που χρειάζεται για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και την προσέγγιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επιπλέον δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών, μεταξύ πυρογνωμών, μεταξύ πολιτών σε διάφορες τομείς όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, αλλά και η καταπολέμηση του εγκλήματος, ε, αλλά και στον πολιτισμό. Και προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με και συνεργασία με τις ε, γειτονικέ χώρες. Έτσι εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθεροποίηση στην περιοχή. Αυτή η ανταλλαγή μεταξύ των λαών, μεταξύ των πολιτών, Χρειάζεται και εμείς αλλά και το Κοσμοπέδιο να προχωρήσουν στην απελευθέρωση από την υποχρέωση ε, θεωρήσεων. Είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου οι πολίτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα. Αισθάνονται εγκλωβισμένοι. Αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά και η απελευθέρωση την υποχρέωση θεωρήσεων πρέπει να γίνει. Του επόμενου μήνε θα ήταν το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λουνατσέκ. Ο Επίτροπος Χάν, εκ μέρους της Επιτροπής, έχει το λόγο. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξότιμα μέλη. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας για την συνεχιζόμενη ανάπτυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοσμοπεδίου. Θέλω να ευχαριστήσω τις Επιτροπές ε, Εξωτερικού Εμπορίου και Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδιαίτερα την εισηγήτρια κυρία Λούνα για τη στήριξη. Αύριο θα ψηφίσουμε τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης την οποία διαπραγματευθήκαμε με το Κωσυφοπαίδιο που είναι ακριβώς η απόδειξη αυτής της ε, πρόοδου. Αυτή η συμφωνία είναι ορόσημο της σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωσυφοπαιδίου και έχει κρίσιμη σημασία για το μέλλον του Κωσυφοπαιδίου και συνολικότερα των Δυτικών Βαλκανίων. Η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη επίσημη συμβατική σχέση που συνδέει την Ένωση με το Κωσυφοπαίδιο και επιτρέπει στο Κωσυφοπαίδιο να συμμετάσχει όπως και η υπόλοιπη περιοχή να, για να απολαμβάνει τα ωφέλη πολιτικά και οικονομικά και να είναι τμήμα της κοινή ευρωπαϊκής προοπτικής που καθιστά την, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ε, ε, ευημερία. Κοινό μας στόχο η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει το κοσφοπέδιο για να κάνει τις ιδιαίτερα αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που θα βασίζονται ε, στο κράτος δικαίων Και έτσι θα δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα που θα δημιουργήσει τη, θέση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα υπάρχει έτσι το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για τη στεδιακή προσέγγιση με τους ευρωπαϊκούς ε, νόμους και προδιαγραφές και θα ευνοήσει και την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, ατόμων και υπηρεσιών και θα ενθαρρύνει χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες του κοσμοπεδίου και θα ενθαρρύνει και την ανάπτυξη του κοσμοπεδίου στον τομέα των μεταφορών και την ενέργεια, γιατί προβλέπει τη σταδιακή ένταξη του κοσμοπεδίου στις ευρωπαϊκές αγορές και την δημιουργία υποδομών ποιότητας. Θα ενισχύσει επίσης την περιφερειακή συνεργασία, διότι το κοσμοπέδιο δεσμεύεται με βάση αυτή τη συμφωνία σε ορατή και βιώσιμη βελτίωση των σχέσεών του με τη Σερβία. Είναι ουσιώδης αρχή της συμφωνίας μας. Η συνέχιση του διαλόγου που διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομική υποχρέωση. Το Κωσυφοπέδιο θα πρέπει να εφαρμόσει τη συμφωνία στην οποία κατέληξε, να συνεχίσει να συνεργάζεται για περαιτέρω συμφωνίες. Όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες, αυτό ορισμένε φορές σημαίνει λήψη δυσχερών αποφάσεων και ανάγκη συμβιβασμών. Τέλος, υπογραμμίζω ότι η συμφωνία περιέχει διατάξεις που δεσμεύουν το κοσμοπέδιο για υψηλού επίπεδου σεβασμό των δημοκρατικών αξιών. Είναι μεγάλες λοιπόν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κοσμοπέδιο. Οι θεσμοί που έχουν δημιουργηθεί για να επιτευχθεί η δημοκρατική διακυβέρνηση και οι κανόνες που επιτρέπουν να λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει καμία παρεμπόδιση του ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου. Η παρεμπόδιση και η βία δεν έχουν καμία θέση σε αυτή τη διαδικασία. Καλό τους πολιτικούς του πεδίου να δεσμευθούν ότι θα υπάρξει ελεύθερη ανταλλαγή πολιτικών απόψεων, ούτω ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, χωρί παρεμποδίσει, χωρίς βία, χωρίς προσπάθειες ε, απειλών και εκφοβισμού. Σας ευχαριστώ για την ε, στήριξή σας και προσβλέπω στην περαιτέρω Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Χάν. Εξ ονόματος Επιτροπής ΙΝΤΑ, ο κύριος Σένφελτ έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να υποστηρίξω την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου. Είναι μια πολύ μικρή χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια και είναι η τελευταία χώρα με την οποία υπογράφουμε μια παρόμοια συμφωνία. Όπως είπε και ο Επίτροπος, αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την μικρή αυτή η χώρα. Ίσως είναι και η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη. Γι' αυτό της προσφέρουμε τη δυνατότητα υποστήριξης και αυτό θα είναι ευεργετικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν λάβουμε υπόψη τη μετανάστευση που αποτελεί ε, μεγάλη πρόκληση για μας, θα μας βοηθήσει και αυτή η χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχουμε τις ομιλητές από τους πολιτικές ομάδες, ο κύριος Αντάκτουσον από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μία συμφωνία ιστορικής σημασίας, διότι η σύνδεση και η σταθεροποίηση με το κοσυφοπέδιο θα αποτελέσει πραγματικότητα. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο ορόσημο για τη χώρα. Έρονται τα προσκόμματα που υπήρχαν μέχρι τώρα και παράλληλα βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι κάτι το δεδομένο. Χρειάζεται πολιτική θέληση και πολιτικές αποφάσεις. Θα πρέπει όμως να γίνουν μεταρρυθμίσεις και βλέπω ότι έγινε λόγος για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό είναι ύψης της σημασίας και αυτό είναι και το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του κοσυφοπεδίου. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εφαρμογή των συμφωνιών κάτι το οποίο επιβάλλεται για να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις και με τις γείτονε χώρες. Είναι κάτι το οποίο αφορά και τις δύο πλευρές. Θα ήθελα να υποστηρίξω λοιπόν αυτή την πρώτη επίσημη συμφωνία που είναι ιστορική. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο εξ των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης με το κοσφοπέδιο προσωπεί ένα βήμα σημαντικό γιατί μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια προώθηση της διαδικασίας ε, γυπνίασης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συμφωνία που εξασφαλίζει συμβατικές σχέσεις με μεγαλύτερο πολιτικό διάλογο, με περαιτέρω εμπορική ολοκλήρωση και νέες μορφές συνεργασίας σε πολυάριθμους τομείς. Φυσικά η συμφωνία είναι σημαντική, αλλά δεν είναι αποφασιστική. Η κατάσταση στο κοσφοπέδιο είναι πολύ προβληματική, όπως είδαμε στις πρόσφατες ε, διαδηλώσεις και η παγίωση της δημοκρατίας και των θεσμών ε, στο κοσφοπέδιο είναι προϋπόθεση για να υπάρχει θετική προοπτική για τη χώρα και για τα Βαλκάνια εν γέννη. Το χρειαζόμαστε κυρίως στη σημερινή φάση που χαρακτηρίζεται από τεράστια προβλήματα, όπως το θέμα της ε, μετανάστευσης και που καθιστούν τα Βαλκάνια και το Σοπέδιο ένα σταυροδρόμι πολύ σημαντικό. Πρέπει να εγκύψουμε επί του θέματος αυτού γιατί μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα από εκεί και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν με την απόλυτη συμφωνία μας ε, και συνένεσή μας αυτή τη συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο παράλληλα να συνοδεύσει το κοσφοπέδιο ε, στην πορεία του. Θα πρέπει η χώρα αυτή να μπει σοβαρά στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της δημοκρατικής σταθεροποίησης και παγιοποίησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κ. Τζαμπάσκι από την ECR. Ευχαριστούμε Είμαστε υπέρ τη συμφωνία σύνδεση και σταθεροποίηση με το κοσφοπέδιο από πλευρά CCR. Χαιρετίζω την προσπάθεια που έκανε η κυρία Λιούνα Σέκα. Το κοσφοπέδιο βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι θεσμοί ε, επηρεάζονται από το πολιτικό βίο, το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί όπω θα έπρεπε, δεν υπάρχει πρόοδος ε, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο ούτε στην καταπολέμηση τη διαφθοράς. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για το κοσμοπέδιο, γιατί χρειάζεται βοήθεια το, η χώρα αυτή για να φτιάξει ένα σύγχρονο κράτος και θεσμούς και για να υπάρξει η οικονομική ανάπτυξη. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη οι, οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων δεν είναι τόσο σημαντικός. Για να μην υπάρχουν ε, εντάσεις και συγκρούσεις θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός όλων των ε, κοινοτήτων, όχι μόνο στο κοσφοπέδιο, αλλά γενικότερα στη χώρα εδώ μιλάω για το φτυφυρό, ε, για, την, ε, για διάφορες μειονότητες ε, που υπάρχουν στα Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντος. Από τους φιλελεύθερους δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, εκ μέρους των φιλελεύθερων θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρως την συμφωνία αυτή με το κοσφοπέδιο. Περιμένω ότι η συμφωνία πλαίσιο επίσης θα υπογραφεί σύντομα για τη συμμετοχή του κοσφοπεδίου στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοσφοπέδιο αντιμετωπίζει αστάθεια σε μια περιοχή που δεν είναι ίδια σταθερή. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Σερβία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχουν αναγνωρίσει τη δημοκρατία του Κοσμοπεδίου. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα ακόμα. Και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δεν επιθυμούν την αναγνώριση αυτού του κράτους και που αναγγέλουν ότι θα αλλάξουν κάποια σύνορα. Αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε σύγκρουση. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας δεν είναι μόνο οικονομική φύσεως συμφωνία. Αφορά την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών, την ενίσχυση της ε, δικαιοσύνης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί πραγματικά αυτή η συμφωνία προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών του Κοσμοπεδίου. Είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι το Κοσμοπέδιο θα, εφαρμο... θα υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η χώρα μπορεί να γίνει και σταθερή και αν γίνει σταθερή θα σταθεροποιηθεί περαιτέρω όλη η περιοχή γιατί είναι τμήμα της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρώπης γεωγραφικά. Γι' αυτό η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να είναι γρήγορη, όσο πιο γρήγορη γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα για μπλε κάρτες απόψε γιατί έχουμε χάσει πολύ χρόνο και θα πρέπει να αρκεστούμε στο χρονοδιάγραμμά μας. Ο κύριος Κόσο για ένα ε, λεπτό. Εμείς ξέρετε ποια είναι η θέση μας για το Κωσυφοπέδιο. Θεωρούμε ότι είναι ένα κράτος που μας έχει επιβληθεί. Γι' αυτό η αυτοαποκαλούμενη δημοκρατία του Κωσυφοπαιδίου δεν συμμετέχει στον ΟΗΕ και δεν αναγνωρίζεται από πολλές χώρες. Σύμφωνα με το ψήφισμα 244 του ΟΗΕ θα πρέπει να αναμείνουμε για μια, σε μια πολιτική συμφωνία και σήμερα η Σερβική Δημοκρατία όπως και η αυτοαποκαλούμενη κυβέρνηση δεν αποτελούν μια πραγματική πολιτική που να διαφοροποιείται από το status quo. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ε, έχουμε να κάνουμε με, μία, ε, ε, με ένα κράτος όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι διάβλοι για να μπορεί να, περνάει, να περνάνε τα, οι Ηνωμένε Πολιτείες τα όπλα τους. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Ζαριανόπουλος. Από τους μη Λόγω της γεωστρατηγικής τους θέσης, δίπλα σε περιοχές που σπαράζονται από ανταγωνισμούς και πολέμους, αποτελούν πέρασμα και προσφύγων αλλά και αγωγών ενέργειας, πεδίο μεγάλων επενδύσεων, προγεφύρωμα της ευρωπαϊκής ένωσης και του νατο σε περιοχές με έντονο ενδιαφέρον και της ρώσικης αστικής τάξης. η πολεμική επέμβαση ευρωπαϊκής ένωσης και νατο έφερε τη διάλυση της ιουγκοσλαβίας έστησε προτεκτοράτα καλλιεργώντας εθνικούς και θρησκευτικούς διχασμούς στους λαούς για την εξυπηρέτηση των ευρωνατοϊκών συμφερόντων και των τοπικών αστικών τάξεων. η συζητούμενη συμφωνία σύνδεσης αναγνωρίζει de facto ένα τέτοιο προτεκτοράτο το κόσοβο έχει τεράστιες ευθύνες και η ελληνική κυβέρνηση που πράττει το ίδιο. πυροδοτεί εθνικισμούς αλυτρωτισμούς μεγαλοδιατισμούς εδαφικές διεκδικήσεις την προώθηση αλλαγής συνόρων όπως η επισήμως απειλούμενη ένωση αλβανίας και κωσόβου σε νέο κράτος με βλέψεις και σε γειτονικές χώρες όπως η φύρομ και η ελλάδα. Ανάλογη αναζωπήρωση εθνικισμών ενισχύει και απαράδεκτη συγκρότηση ομάδα λόμπι ευρωβουλευτών με την ονομασία φίλη τη Μακεδονία. Οι λαοί πρέπει να επαγρυπνούν συμφέρον είναι να αντιπαλέψουν τα υπεριαλιστικά σχέδια να ανατρέψουν τον καπιταλισμό που σπέρνει πολέμους δυστυχία και προσφυγιά. Λοιπόν. Φτάσαμε στην, στο γύρο των ομιλητών. Ε, που μιλούν για λογαριασμό του, ο κύριο Κούκαν. Καταρχά συγχαίρω την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Κοσφοπεδίου που υιοθετούν αυτήν την συμφωνία. Είναι ορόσημο τη σχέσεις μα με το Κοσφοπέδιο το να υπάρξουν συμβατικέ σχέσει. Θα ανοίξει νέε ευκαιρίε για μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοσφοπεδίου. Η συμφωνία δίνει και κίνητρα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη χώρα αυτή είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες περιοχή. Το κοσμοπέδιο θα πρέπει να θεωρήσει ότι η συμφωνία είναι ευκαιρία για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και ευκαιρία για ουσιαστικές πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη για την ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές και τους πολίτες. Η συμφωνία με το Κοσμοπέδιο είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να οδηγήσει εν συνεχεία σε απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων για τους κοσοβάρους. Θα είναι σημαντικό ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και ο λαός του Κοσμοπέδιου να υποφεληθεί πλήρως από τη Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης. Δηλαδή, η Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης είναι βήμα ε, καταργεί εμπόδια στις σχέσεις μας με το κοσμοπέδιο. Θα πρέπει να κάνουμε και άλλα όμως για να χτίσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με το κοσμοπέδιο και το λαό του. Ευχαριστώ. Ο τώρα, και τώρα ο κύριος Πίκουλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Πέδιο σε λιγότερο από ένα χρόνο. Τόσο διήρκεσαν οι διαπραγματεύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αύριο θα ε, επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Έτσι δείχνουμε ότι αναγνωρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική του Κωσυφοπεδίου και προσπαθήσαμε να ορίσουμε συμβατικές σχέσεις και με τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα διότι μπορούμε να προωθήσουμε επενδύσεις, ανάπτυξη και η οικονομική άνοδο αυτής της ε, χώρας, καθώς και ένα κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν ισχύει πάντα κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχει μια τάση παρεμπόδισης αυτής της συνεργασίας που αναγνωρίσαμε τώρα τελευταία, κάτι που δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή πολιτική της χώρας. Εξακολουθούμε να καταπολεμούμε την τρομοκρατία και την ριζοσπαστικοποίηση και θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη συμφωνία μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποτελέσει απαρχή και άλλων μεταρρυθμίσεων. Θα ήταν σκόπιμο το νεότερο ευρωπαϊκό κράτος να τύχει τις υποστήριξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόμασιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου καταβάλει προσπάθειες για την κύρωση αυτής της συμφωνίας. Αυτή είναι η καλύτερη προοπτική, ευρωπαϊκή προοπτική του Κωσυφοπεδίου. Πρόκειται για την νεότερη δημοκρατία στον ευρωπαϊκό χώρο και γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά να ενσωματωθεί στην ευρωατλαντική προοπτική. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για το Πέδιο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής γειτονίας. Ως προς τη διεθνή αναγνώριση θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είμαστε ειλικρινείς υπέρ του κοσυφοπεδίου. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ενώ υπάρχουν χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει τη χώρα. Αυτή η συμφωνία είναι και το πρώτο σημαντικό βήμα για να αναγνωριστεί η χώρα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό καλώ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν το έχουν κάνει και τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Συνατινός έχει το λόγο από τους μη εγγεγραμμένους. Για ένα λεπτό. Το 1999 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έθεσε το Κόσοβο υπό μεταβατική ηγεσία δημιουργώντας κρατήδιο εντός της Ιουγκοσλαβίας και αργότερα της Σερβίας. Το Κόσοβο υπό την ιστορική, γεωγραφική, πνευματική και ηθική πραγματικότητα είναι η καρδιά της Σερβίας και η ψυχή του σερβικού λαού. 17 χρόνια αργότερα και 627 συνολικά από τη μάχη του κωσόβου μεταξύ των ενωμένων σέρβων βόσνιων και κροατών εναντίον των οθωμανών τούρκων η οποία σταμάτησε την προέλασή του στη δυτική ευρώπη κάποια ανιστόρητη και αφελής πολιτική προωθούν τη συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση κωσόβου. αυτό είναι έγκλημα. το κωσόβο δεν είναι κράτος ούτε υφίσταται κωσοβάρικο έθνος. δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εγκλήματα των κομμουνιστών του τίτο που μετάλλαξαν κράτη και βίασαν κυριολεκτικά την ιστορική αλήθεια δημιουργώντας μακεδονικές ονειρώξει και κωσοβάρικα εκτρώματα η προσχώρηση του κωσυφοπεδίου θα αποτελέσει αποδοχή της αλλαγής συνόρων δια της βίας ενός κράτους με μονομερή απόσχεση σερβικού εδάφους βασιζόμενο στα εθνοτικά κίνητρα των αλβανών όπως ακριβώς επιδιώκετε όλοι εσείς να συμβεί με την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της κύπρου. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο είναι ο κύριος Φρουνζουλίκα. Όλες αυτές οι χώρες της ε, Δυτικής Ευρώπης, των Δυτικών Βαλκανίων θα προσχωρήσουν στην Ευρώπη κάποια μέρα. Αυτό είναι κάτι που αφορά και την Ευρώπη και το συμφέρον της. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μογκερίνη για τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Όμως το Βελιγράδι δεν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου και υπάρχουν πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν αναγνωρίσει αυτή τη χώρα. Άρα αυτός ο μηχανισμός είναι ένας μηχανισμός sui για να βρεθεί πιο κοντά το κοσυφοπέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν κάποιον τρόπο ένα τρόπο διαπραγματεύσεων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς την αναγνώριση από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη στάση της Πρίστινας διακόπτεται ο μιλητής από την Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα περνάμε στη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου. Πρώτος είναι ο κύριος Κέλλη. Άκουσα τη συζήτηση είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή συζήτηση. Οι περισσότεροι ήταν υπέρ ε, και κάποιοι κατά αυτής της συμφωνίας. Επειδή είμαι ΕΛΚ, ε, είμαι ιδιαίτερα υπέρ και προσβλέπω στην ανάπτυξη του κοσφοπεδίου και ελπίζω οι κάτοικοί του να έχουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, να αποκτήσουν ιδιαίτερο ε, βιωτικό επίπεδο και ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει περισσότερο εμπόριο και περισσότερη ευημερία. Και προσβλέπω και στη μέρα που θα γίνει το Κοσφοπέδιο πλήρε μέλο τη Ένωση. Είμαι από την άλλη πλευρά τη Ευρώπη. Η Ιρλανδία επίση είναι μικρή χώρα. Στη δυτική πλευρά τη Ευρώπη. Το 1973 γίναμε μέλο τη Ένωση. Και έκτοτε έχουμε αποφεληθεί τρομερά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ούτε θα διανοούμεθα να εγκαταλείψουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και να κάνουν οι φίλοι μα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το νομίζω το ίδιο θα ισχύσει και για το Κωσυφοπέδιο και άλλε χώρε περιοχή. Διότι έχουν πολλά να ωφεληθούν. Πρώτα απ' όλα σταθερότητα, καλύτερε σχέσει γειτονία και φυσικά τι εσωτερικέ μεταρρυθμίσει που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα ο κύριο Σάνι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω, Πρόεδρε. Αυτή η συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην πολιτική γειτονία μας. Η σταθερότητα και η δημοκρατική ανάπτυξη της περιοχής αυτής είναι πολύ σημαντική. Είναι και ώρα να δώσουμε ευκαιρίες στο κοσφοπέδιο καθώς και την προοπτική ταξιδιών χωρίς θεωρήσεις στους πολίτες. Δυστυχώς υπάρχουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναγνωρίζουν το κοσφοπέδιο ως ανεξάρτητο κράτος. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα λοιπόν αυτά τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τη θέση τους που έχει ξεπεραστεί από τις, ε, α, τα γεγονότα. Ο διάλογος μεταξύ Πελιγραδίου και Πριστίνα επίσης είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μπάουτμαντς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Η έκθεση Λούνατσεκ είναι όντως μια έκθεση που αφορά μια πολύ σημαντική συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Θα επιτρέψει το Κοσμοπέδιο να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως. Επίσης, είδαμε και την έκθεση για το τι θα γίνει το 2015 και επιμένω κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι που πρέπει να στηριχθούν, να στηρίξουμε το Κοσμοπέδιο στην οδό αυτήν της πρόοδου και τη προσέγγισης. Ευχαριστώ κύριε Βάουτμαν, ο κύριος Σόλτες. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια κυρία Λούναζεκ για τη θαυμάσια εργασία που έχει πετελέσει, όλες τις προσπάθειες που επένδυσε στα πλαίσια της εκπόνησης αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι η συμφωνία αυτή έχει θεμελιώδη σημασία. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο για το κοσφοπέδιο, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες ε, πέρασε πολύ άσχημες ε, καταστάσεις αυτή η συμφωνία σημαίνει ότι ανοίγει πόρτα για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία και εμπορευμάτων και ατόμων θα διευκολύνει την φλευθεροποίηση των προξενικών θεωρήσεων και φυσικά αυτή η συμφωνία επίσης ανοίγει πολλές δυνατότητες για την ε, ανάπτυξη της ενέργειας, των υποδομών και καθιστά δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που δεν είναι καθόλου αμελητές στο κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι το κοσυφοπαίδιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή. Και αυτό είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφα. Και τελευταίος, ο, και, και τελευταία η συνάδελφος Χολμάιερ στη διαδικασία. Μα δεν είναι μυστικό ότι περισσότεροι ε, πολίτες μας θεωρούν ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη είναι το μαχητικό Ισλάμ. Και αν ε, λάβουμε σοβαρά αυτές τις ανησυχίες ε, του λαού μας, τότε δεν θα δίναμε αυτές τις δυνατότητες στο κοσμοπέδιο. Σήμερα διάβασε μια ελβετική εφημερίδα, στην εφημερίδα Blick, ότι τίθεται το ερώτημα εάν το κοσμοπέδιο θα είναι το πρώτο Ισλαμικό κράτος της Ευρώπης. Και στο άρθρο αυτό τονίζεται ότι οι Σαουδάραβες χρηματοδοτούν την κατασκευή των περισσότερων τζαμιών σε αυτή τη χώρα. Αν θυμάστε, η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα η οποία έχει εφαρμόσει σε πολλές περιπτώσεις βασανιστήρια και έχει καταγγελθεί γι' αυτό. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θεωρεί ότι είναι τέλειος δούριος ύπος στο Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτό το κίνδυνο. Για μένα δεν τίθεται κανένα θέμα γιατί είναι πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε σύνδεση ή ένταξη του κοσμοπεδίου. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Όμπεμάια. Έληξε η διαδικασία προσέλκυση προσοχή του Προέδρου και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χάνη. Χάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπηδίου έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί κλειδί για την Συμφωνία Σύνδεσης και σε ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι μιλάμε για το ίδιο όραμα, την ίδια προοπτική και το ίδιο μέλλον και για αυτή τη χώρα. Μιλάμε λοιπόν για μια ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί μιλάμε για ένα ενδεχομένως, ένα ενδυνάμει μελλοντικό μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να συμμερίζεται τις ίδιες ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή διαχωρισμό μεταξύ θρησκείας και κράτους. Βεβαίως η επόμενη πρόκληση είναι η εφαρμογή. Δεν θα φανούν τα αποτελέσματα άμεσα, θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία όπως συμφωνήθηκε. Δεν πρόκειται για ένα μαγικό ραβδί, δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα, όμως θα νιώσει το κοσυφοπέδιο ότι ανήκει στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιφέρεια και θα δώσει μία πλαισίωση έτσι ώστε το κοσυφοπέδιο να ανταποκριθεί στην ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία όπως επιθυμεί και ο λαός του. Για μία ακόμα φορά θα ήθελα να κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να ε, συζητήσει τις ε, διαφορές με το Βελιγράδι. Δυστυχώς ε, μακρηγορήσαμε και πιστεύω ότι το ψυχοπαίδιο δεν έχει άλλα περιθώρια. Το χρωστάει στο λαό του να βρει λύσεις. Οι πολίτες του Κωσυφοπαίδειου το αξίζουν. Ε, πιστεύω ότι θα είμαι υποστηρίξει το σώμα έτσι ώστε το Κωσυφοπαίδειο να βρεθεί πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Για να κλείσει τη συζήτηση για άλλη μια φορά η συγγήτρια κυρία Λούνατσοκ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επιτροπέ, συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Και, αυτές, και αυτούς που προέρχονται από χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κοσφοπέδιο για την υποστήριξη γενικά που δείχνουν και σε μένα και στη συμφωνία. Ε, θέλω να απαντήσω σε κάποιον που δεν είναι υποστηρικτής ε, ε της Ε, περί πάνω από τα μισά κράτη του ΟΗΕ, 111 έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο. Είναι, είναι και η ώρα να γίνει μέλος του ΟΗΕ το κοσφοπέδιο. Έχουν ακουστεί όλα τα επιχειρήματα. Θέλω να τελειώσω λοιπόν με δύο. Θέλω να επιστρέψω ε, στο, στη μία που έκανα στον Ιμπραήμ Ρουγκόβα. Ε, έτσι ξεκίνησα την παρέμβασή μου σήμερα πρωί. Είναι σύμβολο μια αντίσταση χωριδία. Και θα ήθελα να καλέσω, καλέσω τα κόμματα τη αντιπολίτευση να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ρόγκοβα, να επιστρέψουν ε, στη Βουλή, να, ούτως ώστε να εργαστεί ε, το Κοινοβούλιο, γιατί δεν θα πρέπει σε αυτή τη νέα δημοκρατία να υπάρχει βία στην πολιτική. Και για να τελειώσω, θα ήθελα να πω και κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο είναι καλό για το κοσμοπέδιο. Την περασμένη Πέμπτη, ένα, μια ταινία μικρή ταινία. Ε, από το Κοσμοπέδιο ε, είναι υποψήφια ε, για ένα βραβείο. Λέγεται ΣΟΚ. Ε, μιλάμε για δύο αγοράκια και θα ήθελα αυτό το, αυτή η ταινία μικρού μήκους του Κοσμοπεδίου να πάρει το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία ταινίες μικρού μήκους. Θα είναι μία αναγνώριση για αυτή τη νεαρή χώρα. Ευχαριστώ. Ε, λίγη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο.